την έρευνα. Άρα θα πρέπει να προσέξουμε, δουλεύουμε σωστά όσον αφορά αυτόν τον ε, προϋπολογισμό. Έχουμε εδώ πέρα ένα σωρό προτάσεις, οι οποίες έχουν πάρει το δρόμο τους και θα πρέπει να δούμε τι κάνουμε το 2013. Πώς θα αποκτήσει τα μέσα που χρειάζονται η Ευρώπη. Αλλά αυτό που κυρίως με απασχολεί τι θα γίνει μετά το 2013. Δεν ωφελεί κανείς να ε, ξεκινά με φιλοδοξιδές και να μην μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτές. Θα πρέπει όλοι μαζί να πείσουμε τους ε, πρωθυπουργού, τους ε, αρχηγούς κρατών πώς να έχουν τα μέσα που χρειάζονται. και για τον Τζίμες και για τον Γαλιλαίο. Τι θα κάνουμε. Μέχρι το 2013 θα εγκαταλείψουμε αυτά τα θέματα. Αλλά και ιδίω για το διάστημα θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε το άρθρο 189 θα το αξιοποιήσουμε. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε με την με πολιτική του διαστήματος, ό,τι κάνουμε με άλλες πολιτικές. Έρευνα, καινοτομία, όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε πλήρως. Και άρα έτσι να ξεκινήσει ένα προβληματισμό για να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή πολιτική φιλόδοξη για το διάστημα. Και να δούμε μετά το 2003 πώς θα έχουμε τα απαραίτητα μέσα. Και αυτό να ισχύει και για το Γαλιλαίο, να ισχύει και για το GMS, πολύ για το περιβάλλον, που θέλει η πρόβλεψη δημοσιονομική. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τα θέματα του προπολογισμού. Υπάρχουν ένα πρόβλημα. Δεν μπορούμε να πούμε εντάξει, θα καθαρίσουμε τα τρία πρώτα χρόνια και μετά θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Από τη στιγμή που ξεκινήσουμε προ αυτήν την κατεύθυνση, θα πρέπει να δούμε του τρόπου χρηματοδότηση. Ε, μια, κάποια, ένα καψιλογισμό που θα ήθελα να αναπτύξω εδώ στην Προεδρία, αλλά βέβαια μαζί με το Κοινοβούλιο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πώ θα εντάξουμε, πώ θα διαμορφώσουμε αυτό το 189. Ε, ε, είναι εργασία τη ΕΣΑ βέβαια σε διεθνέ επίπεδο εμεί εργαζόμαστε. Η ΕΖΑ δεν μπορεί να το κάνει αυτό πάντα. Έχει όμω την τεχνική πείρα για την διαχείριση προγραμμάτων και το... η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει πάντα. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να το ψάξουμε αυτό. Τι θα γίνει, πώ θα μπορέσουμε ο ένα να συμπληρώσει τον άλλο και να δούμε και τα κύρια σημεία και των δύο. Ένα να ενισχύσει τον άλλο. Βέβαια και το Βέλγιο θα προσέξει τα πράγματα, αλλά ε, ε, ταυτόχρονα ε, να μην έχει αρνητικέ συνέπειε. Να αποχωρήσει αποχωρήσουν ορισμένα από το πρόγραμμα. Εδώ για τη χώρα μου που γνωρίζω πολύ καλά, από την κυβέρνησή μου το 2008 είχα το 20% του συνολικού ποσού του προπολογισμού για διαστημικά θέματα ακριβώ ε, για το ΕΣΑ ακριβώ και είμαστε από αυτού που συνεισφέρουν ιδιαίτερα. Εντάξει, αλλά τι γίνεται όταν το Βέλγιο επένδυε, Ξέρουμε ότι ο βελγικό ιστό, ο βιομηχανικό, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ξέρουμε τι αντιμετωπίζει μετά, ξέρουμε τα προβλήματα και τον επιχειρησιακό τρόπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, δεν είναι αυτός. Για να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε, πώς θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τα κύρια σημεία, τα ισχυρά σημεία και το με και το δε. Και έτσι να το πετύχουμε αυτό. Και ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός ε, και ο διαστημικός χώρος να παραμείνει αντικείμενο και προσοχής και να δούμε είναι κάτι που θα πρέπει να το προσέξουμε σίγουρα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και στις 21 Οκτωβρίου θα δούμε για την εξέμβαση του διαστήματος. Ο κ. Ομπαμά θα συμμετάσχει και η Κίνα και η Ρωσία επίσης ιδιαίτερα ενδιαφέρονται. Είναι ε, στα starting block πάνω σε αυτό και θα πρέπει να δούμε τι θα κάνει η Ευρώπη, πώς θα μπορούσε να συμμετάσχει για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε. Γιατί η Ευρώπη όταν συμμετέχει εκεί το κάνει με δύο τρόπο. Σας μίλησα και την Ευρώπη και βέβαια αυτό που μας απασχολεί πάντα είναι ε, όσο γίνεται περισσότεροι και η Αφρική μηχανή που δεν μπορούν να μείνουν ε, στην άκρη, στο περιθώριο. Πώς θα μπορούσαν να μετάσχουν οι περισσότεροι για ευμάρεια του πολίτη, για τη χρήση αυτού του διαστήματος και αυτή είναι η φιλοδοξία σε παραμεδιαστημικά θέματα, η φιλοδοξία του Βελγίου. Για μικρομεσαίε επιχειρήσεις δεν ξέρω τι να σας πω. Εντάξει, θα πρέπει να πούμε, υπάρχουν αρκετοί από εσά που έρχονται από μεγάλες χώρες ε, και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι διαφορετική άποψη περί μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και τώρα ε, το 99,9% 10% των επιχειρήσεων των βελγικών είναι με 250 άτομα, αν πάρουμε αυτόν τον αριθμό. Εντάξει, θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν μιλάμε για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, το ίδιο πράγμα δεν εννοούμε. Πάντως, ε, αρκετά σημαντικά μέτρα πήραμε ε, και μειώντας τη φορολογία των ε, ερευνητών ε, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει κατά τη διάρκεια προεδρίας μας, πώς αυτό το Small Business Act να οδρεωθεί περισσότερο στα κράτη-μέλη μας και τι θα κάνουμε να μην έχουμε το ίδιο πράγμα, να μιλάμε για το ίδιο πράγμα αλλά είναι διαφορετικό, θα πρέπει να συμμεριστούμε και να μοιράσουμε την πείρα μας. Πρέπει να δούμε πώς θα απλοποιήσουμε για τη επιχειρήσει επιχειρήσεις, υπευθυνοί τους, πώς οικονομική δραστηριότητά τους να αναπτυχθούν, ταυτόχρονα όμως να είναι καρφωμένοι στο ίντερνετ, μήπως υπάρχει κάποιο υποεδάφιο που τους απασχολεί και τους ενδιαφέρει. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι μπορούμε να κάνουμε. Εδώ θα πρέπει να δούμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να δούμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα έρευνα σε μικρομεσαίο, σε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι δεν το κάνουν τελικά, το χρησιμοποιούν επειδή δεν έχουν τον χρόνο, επειδή δεν ξέρουν γίνεται κλπ. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν συμμετέχουν λοιπόν σε αυτή την ανάκαμψη την οικονομική, να συμμετάσχουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και με πρόσβαση στην καινοτομία. Ο τρόπο είναι απλοποίηση, απλοποίηση, απλοποίηση. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα προσπαθήσω να απαντήσω στι ερωτήσει όπως ετέθησαν και να μην επαναλάβω πολλά πράγματα. Κύριε Καρβάγιο, σωστά είπε κάποια πράγματα για το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε, τα κονδύλια της υπαίθρου για την ευρυζωνικότητα. Κοιτάξτε, θα καταθέσει η Κομισιόν την πρόταση της για τη στρατηγική της ευρυζωνικότητας και είπε πως πρέπει να τα δούμε τα πράγματα αντίστροφα. Αντί να βλέπουμε τα διαρθρωτικά, τα μία μεμονωμένα, τα δούμε σε μια ευρύτερη ε, στρατηγική. Αυτό νομίζω πολύ σημαντικό και πολύ θετικό. Δεύτερον, η Κομισιόν θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη για να δουν τι μπορούν να κάνουν με την υβριζονικότητα μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν όσο δυνατόν περισσότερο αυτά τα κονδύλια. Γιατί το κόστος για τους φιλόδοξους αυτούς στόχους που έχουμε για 2013 και 2020 μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που είτε θα πρέπει να τα δώσουν ιδιωτικές επιχειρήσεις ή τα κράτη ε, αλλά ξέρετε πως αυτό είναι δύσκολο αλλά θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αυτά προβλέπονται στο σχέδιο ανάκαμψης της Ευρώπης αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ΣΔΙΤ σε ιδιωτικό τομέα να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν στο μαγίστο τα κονδύλια δεύτερον το ερώτημα του κυρίου Ρούμπιχ για το roaming, την περιαγωγή. Ο κύριος Ρούμπιχ μίλησε για το LTE, τα δίκτυα τέταρτης γενεάς, τα οποία μπορούμε να καταργήσουμε το roaming απευθείας. Έχουμε το ψηφιακό σχέδιο της κυρίας Κρούς για να φτάσουμε μέχρι το 2015 σε ένα ΣΕΤΑ. Έχουμε το λεγόμενο ΣΕΤΑ, δηλαδή τον ενιαίο χώρο πληρωμών και να έχουμε και τον ενιαίο χώρο τηλεπικοινωνιών. Οπότε να μην έχει σημασία από πού ξεκινάει κανείς, αλλά να κινείται σε μια τηλεπικοινωνιακή ευρωζώνη και να υπάρχει μια ενιαία χρέωση επαναστατική ιδέα και απαραίτητη. Το 2015 μου μοιάζει και κάπως αργά. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι. Για να δούμε τι θα κάνουμε με το LTE. Ίσως ευθύς εξ αρχής καλά τα λέτε. Καλή ιδέα. Νομίζω πως πρέπει λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιδείξει εδώ πέρα αυτοπεποίθηση. Να προτείνει ένα κείμενο πει, ε, δεν ξέρω, ένα ψήφισμα, δεν ξέρω πώς ε, τα λέτε αυτά εδώ πέρα. Να το στείλει στην Κομισιόν και, η Προεδρία, και στην Προεδρία μας και η Προεδρία θα βρει έναν τρόπο. Ε, η κυρία Φιγκορέδο είπε πως υπάρχουν και άνθρωποι στις πόλεις που χρειάζονται ευρυζωνικότητα. Μιλήσατε για ένα 20% παραδείγματο χάρη ε, πως ε, στο Βέλγιο ε, μόνο ένα 70% είναι συνδεδεμένο σε ευρυζωνικότητα και ξέρετε πως άρα ένα 30% δεν είναι συνδεδεμένο, έχει προβλήματα, άρα δεν μπορεί π.χ. να κάνει τραπεζικές συναλλαγέ μέσω ίντερνετ. Οπότε θα πρέπει να δούμε αυτή τη συζήτηση για το αν πραγματικά υπάρχει, ε, αν θα το καταστήσουμε αυτό μια καθολική υπηρεσία η οποία θα πρέπει να παρέχεται. Θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, ως ε, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θεωρούμε εμείς ε, πως θα πρέπει το ευρυζωνικό ίντερνετ να είναι μια καθολική υπηρεσία Πράγματι είναι ένα βασικό δικαίωμα, όπως είπατε κι εσείς, ε, είναι νομίζω συγκρίσιμο με άλλες βασικές υπηρεσίες και μπορεί να περάσει στις, στην καθολική υπαρχή. Κυρία Τόμψεν αναφέρθηκε σε κινδύνους για την υγεία. Ξέρετε πως ούτως ή άλλως το πλαίσιο το θέτει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, και σωστό αυτό το οποίο λέει το Ινστιτούτο Στοκχόλμη, ε, θα δούμε τώρα. Γνωρίζουμε τους πιθανούς κινδύνους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, έτσι. Γιατί εμφανίστηκε μια έκθεση στη Γαλλία για πιθανούς ε, κινδύνους υγείας και γνωρίζω πως η κυρία Κρούς ε, έχει μια σχετική στρατηγική, γνωρίζω το, το πρόβλημα, αλλά δεν πρέπει να το βλέπουμε ιδεολογικά, α, παρά μόνο επιστημονικά. Η κυρία Φανμπρέντ μίλησε για το roaming πάλι δεδομένων. Ξέρετε, ήταν σαφές το 10 στις 8 Ιουνίου. Είπε δηλαδή πως οι εδρεωμένες εταιρείες ε, οι απόλυτα λαμβάνουν κάποια προνόμια και Πράγματι εδώ πέρα βλέπετε ότι δεν είναι διαφανής καθόλου η αγορά της περιεγωγής για να μπορεί να κάνει επιλογές ο καταναλωτής. Εάν δει κανείς τις τεράστιες διαφορές μεταξύ κλήσεων και δεδομένων εσωτερικού και εξωτερικού αναρωτιέται μα τι δεν δουλεύει εδώ πέρα. Πρέπει λοιπόν πράγματι να δείξει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Βεβαίω να ακολουθήσουμε την απόφαση του ΔΕΚ και όταν καταθέσει την πρότασή της η Κομισιόν να πάει περισσότερο στην κατεύθυνση νομίζω ε, ανώτατων τιμών και να μην περιμένουμε άλλο γιατί κάθε καλοκαίρι περιμένουμε και βλέπετε τι, τι γίνεται. Ξέρετε πως υπάρχει μια ειδοποίηση όταν φτάσει κανείς στα 50 ευρώ, αλλά νομίζω πως δεν επαρκεί κάτι τέτοιο. Και Για το ΕΝΖΕ βέβαια επιτέλους είναι ώρα να μας έρθει η Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις μέσα σε Επτεμβρίου κανονικά επιτάπητος θα πρέπει να θέσει και προτάσεις και τα εργαλεία για να πετύχουμε αυτή την ισορροπία και ίσως joint ventures για ώστε οι διάφοροι φορείς να ξεύρουν τα χρήματα και να έχουν και την δυνατότητα το FTTH να αναπτύξουν. Μιλάμε για δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Α, λοιπόν, ε, δεν θα πρέπει να έχουμε βαλίσει, θα είναι σημαντικότατη επένδυση Ίσως δεν υπάρχει αρκετός ανταγωνισμός, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε για ένα άνοιγμα ή για μια λογική συμτιμή και για άλλους ανταγωνιστές. Ε, αυτά ήθελα να... Και θα ολοκληρώσω κύριε Πρόεδρε γι' αυτό. Η θέση του Κοινοβουλίου κανονικά, αν θυμάμαι καλά, το Μάρτιο φέτος ε, ότι απαιτείται διαφάνεια. Αυτό θα πρέπει να γίνει σεβαστό. Και τι κάνουμε τώρα. Ολοκληρώνουμε τη φάση αυτή. Έχουμε ακόμα στο τέλος του μήνα αυτή μια συνάντηση στο Τόκιο και υπό την Βελική Προεδρία αυτό το άκτα θα ολοκληρωθεί, θα περατωθεί, θα πρέπει να επιμείνουμε πάντα για μια διαφιόνια Έστω και αν ακούμε φήμες από τη μια ή την άλλη πλευρά, αλλά και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σας εξήγησε τη θέση του ΑΚΤΑ εδώ μπροστά σας. Χρειάζεται να σεβαστούμε και άλλες ισορροπίες όπως την 138 τροπολογία και αυτό που τη δίδεται στα πλαίσια του Telecom Package. Πετύχαμε, θα πρέπει να το προσέξουμε και καταλαβαίνουμε ότι απαιτείται απόλυτη διαφάνεια. Μην μπλέξουμε σε περιπέτειες τώρα που δεν επιθυμούμε έτσι και δεν θα υπάρχει καμία λύση και θα μπορούσαν να συνδυαστούν όλα αυτά τα πράγματα με ό,τι έχει ήδη αποφασίσει η Ευρώπη και βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά κύριε Πρόεδρε, ολοκλήρωσα. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ τους Υπουργούς πρώτα απ' όλα για τις συνθήκες υπό τις οποίες συνομιλήσαν μαζί μας. Δεύτερον, ευχαριστώ τους διερμηνείς ε, που παρέμειναν λίγο παραπάνω. Και τρίτον, θα περάσουμε στα διάφορα. Στην αρχή της συνεδρίασης είπαμε πως θα πρέπει να δούμε το ερώτημα της ε, Επιτροπής Περιβάλλοντος για την COP16. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, νομίζω μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ τα